Συνάδελφοι, δεν έχουν προσελθεί όλοι ακόμη. Παρ' όλα αυτά θα πρότεινα να ξεκινήσουμε. Σας καλωσορίζω στην ε, σημερινή μας συνεδρίαση όλους και ξεκινώ με την έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης. Δυστυχώς πρέπει να σας ενημερώσω ότι η κυρία Αζουλάη, η Γενική Διευθύντρια της UNESCO, ε, ήταν αναγκασμένη να ματαιώσει τη σημερινή μας συνάντηση. Θα προσπαθήσουμε όμως να ορίσουμε νέα ημερομηνία το συντομότερο δυνατό. Αυτό σημαίνει ότι το απόγευμα θα γίνει η συζήτηση με την Κομισιόν για την αξιολόγηση του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη. Ε, θα γίνει νωρίτερα, δηλαδή ακριβώς στις 3 το απόγευμα. Λοιπόν, εγκρίνεται η σε διάταξη με την τροποποίηση αυτή. Χέλγα. Θέλω να εξασφαλίσουμε ότι η κυρία Ζουλάη θα έρθει το συντομότερο δυνατό. Θα προσπαθήσουμε και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, είπε η Πρόεδρος. Ήταν προσκεκλημένη, ε, είχε επιβεβαιώσει την παρουσία της. Προχθές μόλις μας ενημέρωσε ότι τελικά δεν θα τα καταφέρει να βρίσκεται εδώ. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να ε, ορίσουμε νέα ημερομηνία το συντομότερο δυνατό. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Αλλά όπως είπα θα προσπαθήσουμε να ορίσουμε νέα ημερομηνία. Λοιπόν, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίρρηση σχετικά με τη μίληση διάταξη. Επομένως εγκρίνεται. Περνάμε στο δεύτερο σημείο της ημίλησης διάταξης, έγκριση των πρακτικών το σχέδιο πρακτικών των συνεδριάσεων της 19ης και 20ης Μαρτίου τα έχετε λάβει στα έγγραφά σας. Έχετε κάποιες παρατηρήσεις ενδεχομένως να κάνετε για τα πρακτικά. Όχι από ό,τι βλέπω. Επομένως θα πρότεινα ως συνήθως να θεωρήσουμε ότι τα πρακτικά έχουν εγκριθεί εφόσον δεν υποβληθούν αντιρρήσεις, ενστάσεις στο τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Ανακοινώσεις Προέδρου. Καταρχάς, να καλωσορίσω μια νέα σύμβουλο της πολιτικής ομάδας, την Άννα Γκόρνη, για την ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Επίσης, υπάρχει διερμηνία για τις εξής γλώσσες, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εσθονικά, ουγγρικά, πολωνικά, βουλγαρικά και ρουμανικά. Να σας υπενθυμίσω όπως πάντοτε ότι η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο και οι αποφάσεις των συντονιστών της 25ης Απριλίου 2018 Μπορώ να σας ενημερώσω ότι οι αποφάσεις των συντονιστών της ημέρας αυτής που απεστάλησαν σε εσά τα μέλη της Επιτροπής Κούλς στις 26 Απριλίου έχουν εγκριθεί επισήμως καθώς μέχρι τις 30 Απριλίου που ήταν η προθεσμία Α, όχι, συγγνώμη, όχι, συγγνώμη. Υποβλήθηκαν δύο παρατηρήσεις σε σχέση με αυτές τις αποφάσεις σχετικά με το προφορικό ερώτημα της, προ... της Επιτροπής Πέτη. Δεν επηρέαζαν άμεσα βεβαίω τις αποφάσεις των συντονιστών. Παρ' όλα αυτά, σήμερα στη συνεδρίε των συντονιστών θα ξανασυζητήσουμε αυτό το αίτημα τη Επιτροπής πέτη, το έχουμε ξαναβάλει στην σε διάταξη. Αλλά, όπως είπα, δεν επηρεάζονται οι ίδιες οι αποφάσεις των συντονιστών, επομένως ε, θεωρούν ότι έχουν εγκριθεί. Εφόσον δεν ε, λάβαμε επί της ουσίας παρατηρήσεις. Και μπορούμε να περάσουμε απευθείας στην ψηφοφορία. Ψηφοφορία για σχέδιο γνωμοδότησης σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία βάσει του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17 η Μαΐου 2017. Συντάκτρια της γνωμοδότησης είμαι εγώ. 76 τροπολογίες λάβαμε. Έχω προτείνει 10 συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ όλους τους σκιώδεις εισηγητές για την επικοδομητική μας συνεργασία. Για αυτό το πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου θέμα και νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Να βρω λίγο την κάρτα μου. Βρείτε την κι εσείς ο καθένας. Ζητώ συγγνώμη και ξεκινάμε απευθείας. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε με την συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 5. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε παρακαλώ πέρας εφορία εγκρίνεται 13 υπέρ 11 κατά και περνάμε στην τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ναι, αν θέλετε μπορούμε να το ελέγξουμε. Ναι, θέλετε να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, βεβαίως. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά επί της τροπολογίας 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 9 υπέρ 14 κατά. Τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ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 Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 και 55 που ταυτίζονται υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 61 υπέρ, κατά,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 κατά αποχές εγκρίνεται. 74 με προφορική ε, τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 75 υπέρ Θέλετε να το ελέγξουμε. Εντάξει, να ελέγξουμε την 74 με την προφορική τροπολογία. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά άρχη ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 14 υπέρ, 11 κατά. 75 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να το ελέγξουμε να είμαστε σίγουροι. Ξεκινάει λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 76. Πέρας. Ναι, πράγματι. Ήταν μικρή η διαφορά. 12 υπέρ, 13 κατά, άρα απορρίπτεται. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία που θα γίνει ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ επί του συνόλου τη γνωμοδότησης. Geschlossen. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 13 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 8 αποχές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. και περνάμε στην επόμενη, στο επόμενο σημείο της υπηρεσίας διάταξης εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης για την ενίσχυση της ανάπτυξης και της συνεργασίας σε μεθοριακές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγγητής είναι ο συνάδελφος Ζαγοράκης. στον οποίο και δίνω το λόγο. Το πολύ για πέντε λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η προώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής στι παραμεθόρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και νομίζω ότι σωστά η Επιτροπή μας κλήθηκε να γνωμοδοτήσει επί του θέματος. Οι εσωτερικές παραμεθόρες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιπροσωπεύουν το 40% της επικρατείας και φιλοξενούν 150 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Παρ' όλα αυτά, οι οικονομικές τους επιδόσεις υπολείπονται σημαντικά των άλλων περιφερειών στο εσωτερικό των κρατών μελών. Εμπόδια κυρίω διοικητικά αλλά και νομικά παρεμποδίζουν την ανάπτυξη και τη συνοχή στι παραμεθόρειε περιφέρειες. Οφείλουμε να δράσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχοντα ωστόσο στοχευμένη προσέγγιση για κάθε περιοχή ξεχωριστά. Το θέμα έχει πολλές προεκτάσεις, αλλά θα επιμείνω στο κομμάτι που άπτει των αρμοδιοτήτων της δικής μας Επιτροπής. Αγαπητοί συνάδελφοι, το πιο σημαντικό για μένα είναι να υπάρξει απαραίτητη πολιτική βούληση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταφέρουμε να μεταδώσουμε το αίσθημα της εμπιστοσύνης που απαιτείται σε τέτοιου είδους εγχειρήματα. Ο πολιτισμός, η παιδεία και ο αθλητισμός αποτελούν προνομιακό πεδίο προς αυτή την κατεύθυνση. Γι' αυτό το λόγο <clears throat> πρέπει να το εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Τα προγράμματα αυτά μπορούν να φέρουν τους Ευρωπαίους πολίτες πιο κοντά και να βοηθήσουν στην οικονομική ανάπαξη των παραμεθόρων περιφερειών. Ο μεγάλος αριθμός σχεδίων Interreg είναι, που είναι αφιερωμένα στον πολιτισμό αποδεικνύει ότι υπάρχει έντονη επιθυμία μεταξύ των παραμεθορίων περιφερειών να επενδύσουν σε κοινά πολιτιστικά project και γι' αυτό το λόγο πρέπει να στηρίξουμε ουσιαστικά τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες στα πλαίσια του επόμενου πολιετούς δημοσιοοικονομικού πλαισίου. Παράλληλα, η συστηματική προώθηση της πολυγλωσία στην εκπαίδευση αλλά και την επαγγελματική κατάρτιση στι παραμεθόρειε περιφέρειε μπορεί να αποτελέσει τη λύση σε πολλά προβλήματα που παρουσιάζονται στα σχέδια διασυνδρομική συνεργασίας. Τέλος, τα κράτη-μέλη μπορούν και οφείλουν να, να διευκολύνουν και να ενθαρρύνουν την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μεταξύ των γειτονικών περιοχών. Η προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει. Παρ' όλα αυτά, παραμένουν ακόμη πολλά γραφειοκρατικά προβλήματα που πρέπει να επιληθούν το συντομότερο δυνατό. Δεν θέλω όμω να μακρηγορήσω. Προτιμώ να ακούσω τι απόψει συναδέλφων από τι άλλε πολιτικέ ομάδε. Είμαι πραγματικά ανοιχτό στα σχόλια και στι παρατηρήσει του. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μπορούμε να βρούμε κοινή συνισταμένη και να καταλήξουμε σε ένα κείμενο με ευρεία συνένεση. Λόγω των περιορισμών στην έκταση του κειμένου περιορίστηκα στα απολύτω απαραίτητα. Γι' αυτό το λόγο θα καταθέσω και εγώ κάποιε τοπολογίε όπου θα, εξειδικευ... θα εξειδικεύω ορισμένα σημεία στα οποία έπρεπε να είμαι πιο περιεκτικό. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ζαγοράκη. Ας ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις εισηγητές. κυρία Μίτση, το πολύ τρία λεπτά σας παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε τις τελευταίες ε, δεκαετίες η ευρωπαϊκή διαδικασία ολοκλήρωση έχει βοηθήσει τις παραμεθόριες περιοχές να μετατραπούν από περιφερειακές και απομακρυσμένες περιοχές σε περιοχές ε, Ευημερία. Βεβαίω έχουν μεγαλύτερε προκλήσει να αντιμετωπίσουν από τι υπόλοιπε ευρωπαϊκέ περιοχέ και έτσι η συνεργασία μεταξύ, διασυνοριακά μεταξύ των περιφερειών αυτών ε, βοηθά πολύ στην αντιμετώπιση και προσκομμάτων αλλά και στον περιορισμό των δυσμενών συνθήκων που ως εκ τους ε, αντιμετωπίζουν και βεβαίως μπορεί να οδηγήσει και στη βελτίωση των συνθήκων για την ε, ολοκλήρωση, συνεργασία, εκπαίδευση, αθλητισμό κτλ. Το πρόγραμμα Interreg έχει ιδιαίτερα βοηθήσει τις περιοχές αυτές να μεταμορφωθούν. Προγράμματα συνεργασίας έχουν συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομίας της στηριζόμενης στη γνώση, να ενισχύσουν στην ενίσχυση των επενδύσεων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων μέσα στις τοπικές οικονομίες. οικονομίες. Βεβαίως υπάρχουν τεχνικά, νομοτεχνικά και κανονιστικά προβλήματα και εμπόδια που εμποδίζουν την ανάπτυξη αυτών των περιφερειών εις βάρος της ε, ελεύθερης ε, κίνησης ε, πολιτών πρώτα απ' όλα κεφαλαίων, ιδεών, εμπορευμάτων. Πρέπει λοιπόν να ενισχυθεί αυτή η κινητικότητα. Η πολιτική της συνοχής στις παραμεθόριες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απαραίτητη για να συνεχιστεί η προσπάθεια για την ενίσχυση της ενίσχυσης ε, με την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση που δίνεται για τη ε, συνοχή από τη μία πλευρά των σύνορων οπωσδήποτε θα αντανακλάται και από την άλλη πλευρά. Και γι' αυτό καλωσορίζω την έκθεση του κυρίου Ζαγοράκη, η οποία είναι ένα ε, εξαιρετικό σημείο κίνηση για τη συζήτησή μα. Ω εισηγητή, κατάφερε να καταγράψει τα πιο σημαντικά σημεία στα προγράμματα διασυνοριακή συνεργασία και ιδιαίτερα σε ζητήματα εμ χρηματοδότησης του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του αθλητισμού που αφορούν τους πολίτες, αλλά και άλλα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες πέραν των σύνορων και πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί ε, πάντα ε, χρηματοδοτική υποστήριξη στα πολιτιστικά έργα, ιδιαίτερα με έμφαση στην πολυγλωσία, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση, ο, ο μεταξύ, η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και τεχνικών ιδρυμάτων, τεχνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Η συνεργασία ωστόσο πιστεύω πρέπει να ξεκινά από, το, από τα πρώτα χρόνια τη ηλικία. Να υπάρχουν διασυνοριακέ ανταλλαγέ σχολικέ επισκέψει, δηλαδή, να γνωρίζουν τα παιδιά το ένα το άλλο ακόμα και σε αυτή την ε, μικρή ηλικία του δημοτικού πέραν των συνόρων για να απελευθερωθεί το δυναμικό των ε, νεαρών παιδιών πέραν των σύνορων. Έχουν τη δυνατότητα τα παιδιά νομίζω να αξιολογούν και να καταλαβαίνουν την ποικιλία, την διαφορά, την πολυγλωσία, την ε, πολιτιστική πολυμορφία. Μέτρα αντίστοιχα ε, άλλα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν όπως ερευνητικά κέντρα, κέντρα συνεργασίας εκπαιδευτικά κτλ. Και έτσι μπορεί να περιοριστεί και η φτώχεια και η ανεργία της νεολαίας και ο κοινωνικός αποκλεισμός στις περιοχές αυτές. Έτσι λοιπόν είναι αυτά τα περιφερειακά έργα τεράστια σημασία για την νεολαία και ακόμη περισσότερο για την Επιτροπή μας, για την πέραν των αρμοδιτών δηλαδή τη Επιτροπή μα, έχουν τεράστια σημασία για την οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των περιφερειών αυτών. Σα ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Η κυρία Evans. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εισηγητή για το σχέδιο γνωμοδότησης, για τη σημασία της ε, εκπαίδευσης του πολιτισμού, του αθλητισμού σε τέτοια έργα. Εγώ εκπροσωπώ την ε, ε, Ουαλία με εξαιρετικές εμπειρίες σε σχέση με υπερσυνοριακά προγράμματα, ιδιαίτερα στην Ιρλανδία. Ξέρουμε πόσο πολύτιμα είναι για τον πολίτη. Είναι ε, προγράμματα επαφής πολίτη με πολίτη, ανθρώπου με ανθρώπου και αυτό είναι η μεγάλη τους δύναμη. Νομίζω ότι η γνωμοδότηση καλύπτει όλα τα σημαντικά σημεία. Με ικανοποίηση βλέπω ότι υπάρχει παραπομπή στη γλώσσα, τους γλωσσικούς φραγμούς, τη σημασία της τεχνολογίας της γλωσσικής που θα μπορούσε να βοηθήσει να υπερβληθούν ε, οι φραγμοί αυτοί. Ε, πολύ σημαντικό το ότι υπογραμμίζεται. Αθλητισμός, πολιτισμός, τουρισμός, όλα αυτά πολύ σημαντικά για τις εκλογικές μας περιφέρειες. Η, ο κλάδος του πολιτισμού, ο κλάδος της καλλιτεχνικής δημιουργίας έχει τεράστια σημασία, ιδιαίτερα για τη δική μου την περιοχή, την Ουαλία. Και θα ήθελα ιδιαίτερως να εξετάσω δυνατότητες για ενίσχυση και υποστήριξη και της περαιτέρω συνεργασίας. Βεβαίως για μας είναι κάπως αβέβαιες οι εποχές και έτσι η δυνατότητα για διαφύλαξη της ελεύθερης κυκλοφορίας και διακίνησης πέραν των συνόρων θα έχει τεράστια σημασία για τον πολιτιστικό τομέα και την καλλιτεχνική δημιουργία στην περιοχή μας. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και να προσπαθήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, υπογραμμίζοντας ελπίζω και μέσα στο κείμενο ε, τη διάσταση αυτή. Ευχαριστώ. Κυρία Καμερέβερτ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σχοντής. Τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Ζαγοράκη, για την γνωμοδότηση, την οποία θεωρώ πολύ εύστοχη, γιατί δεν είναι εύκολη δουλειά. Μέσα σε λίγα, λίγες λέξεις, λίγες φράσεις που περιορίζει η γνωμοδότηση, να θίξει ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και κατά τη δική μου άποψη. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να πω ότι σας είναι γνωστό, το έχουμε διαπιστώσει, ότι δυστυχώς το τελευταίο διάστημα ε, έχουν ενισχυθεί οι κοινωνικές αλλά και περιφερειακές ανισότητες στην Ευρώπη και θύμα αυτής της διεύρυνσης των περιφερειακών ανισοτήτων, τουλάχιστον με βάση τη δική μου εμπειρία από την Ελλάδα, δηλαδή οι πιο υποβαθμισμένες είναι οι παραμεθόριες. παραμεθόριες. Οι λόγοι είναι συγκεκριμένοι, δεν θα τους αναλύσω τώρα. Επομένως υπάρχει ένα θέμα να ενισχυθούν οι παραμεθόριες περιοχές και από την άποψη της ανάπτυξης και από την άποψη της συνοχής. Η δεύτερη παρατήρηση που θέλω να κάνω, συνήθως όταν θίγεται αυτό το θέμα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, προσανατολίζεται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο η τον αλλο τροπο πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των εμπορικών και των οικονομικών ανταλλαγών. Στο όνομα των ελευθεριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ούτω καθεξής. Καλός, κακός είναι μια συζήτηση. Καλός λέω. Αυτά όμως από μόνα τους δεν επιφέρουν βήματα συνοχής και ανάπτυξης του τομεί με του οποίου ασχολείται η Επιτροπή μας. Δηλαδή η παιδεία και ο πολιτισμός δεν προκύπτει επειδή θα αναπτύξεις περισσότερο τις οικονομικές ανταλλαγές. Γι' αυτό συμφωνώ με τον εισηγητή ότι χρειάζεται και πολιτική βούληση, χρειάζεται και σχεδιασμός. Δεν προκύπτει, επαναλαμβάνω από μόνα του, σύμφωνα με ένα σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης θα μας προκύψουν ε, προθυμένα βήματα στη συνεργασία και σε αυτούς τους τομείς που θέλουν μια ιδιαίτερη φροντίδα, μια ιδιαίτερη προτεραιότητα και με αυτή την έννοια συμφωνώ, ξαναλέω με τον εισηγητή, ότι θέλει πολιτική βούληση μεν, θέλει και συγκεκριμένε προτάσει, προγράμματα, σχεδιασμού, συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να το πετύχουμε. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, ε, βλέπω τι προτάσει που κάνει ο εισηγητή, ε, θα τι μελετήσω καλύτερα, θα τι μελετήσουμε καλύτερα και θα καταθέσουμε τι σχετικέ τροπολογίε. Και πάλι ευχαριστώ τον εισηγητή, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα συμβάλλουμε και εμεί ώστε να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρία Σόντροβα, παρακαλώ, δύο λεπτά. Ε, ε, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον χρωμοδότη για την πολύ καλή γνωμοδότηση, το ρόλο του πολιτισμού που έχει εξάρει ιδιαίτερο. Εγώ προέρχομαι ίδια από περιφερειακή, από παραμεθόρια περιφέρεια και είναι πάρα πολύ σημαντικό πιστεύω να τονιστεί ότι είναι μεγάλος ο κίνδυνος να εγκαταλείψουν οι πολίτες, όπως ήδη συμβαίνει τις περιοχές αυτές. Βλέπουμε μια απερίμωση των περιοχών αυτών. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία να αναπτύξουμε εκείνες τις δραστηριότητες που θα επιτρέψουν στον πολίτη ή να μείνει στην περιοχή ή να επιστρέψει. Σε αυτό πρέπει ιδιαίτερα να στοχεύσουμε, δηλαδή να αποφύγουμε, να σταματήσουμε την εγκατάλειψη από τους πολίτες αυτών των περιεχών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Φερχάιεν. Ναι, είναι λίγος ο χρόνος, δύο λεπτά μόλις από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν ε, θα επεκταθώ λοιπόν στο πρόγραμμα Interreg. Νομίζω ότι ο τίτλος «Προαγωγή και ανάπτυξη στις παραμεθόριες περιοχές», ο τίτλος όπως έχει καταγραφεί νομίζω είναι ιδιαίτερα σημαντικός και ξεκάθαρος και εγώ προέρχομαι από περιφερειακή, από παραμεθόρια περιοχή και Νομίζω ότι πρέπει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού ε, από το γειτονικό Βέλγιο, το γερμανόφωνο, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναγνωρίζεται χωρίς ε, ναι μεν αλλά και υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα στα οποία μπορούμε να ε, συνεργαστούμε. Βεβαίως μπορεί να βοηθήσει το Interreg, αλλά οτιδήποτε κάνουμε με ό,τι ρυθμίσεις θα πρέπει να επιδιώκει τη μεγαλύτερη ευελιξία και κινητικότητα πέραν των σύνορων. Ελευθερία, κινητικότητα, ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, ελεύθερη διακίνηση υπηρεσιών, εμπορευμάτων. Αυτά πρέπει να ε, βοηθήσουν για να αναζωογονηθούν οι περιοχές αυτές και να απαλληφθούν οι ε, φραγμή. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή εγώ που ζω σε μια παραμεθόρια περιοχή να πάω ή να στείλω το παιδί μου στο σχολείο της γειτονική χώρας πάλι στην παραμεθόρια περιοχή. Αυτά τα πράγματα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πάντως είναι πολύ καλή γνωμοδότηση και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λιμπάτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετίζω και εγώ ε, την προσέγγιση του εισηγητή. Θέλω όμως να τονίσω και την πολιτική σημασία που έχουν οι παραμεθόριες περιοχές. Διότι οι παραμεθόριες περιοχές είναι, πώς να σας πω, η βιτρίνα της Ευρώπης σε πάρα πολλές χώρες. Και γι' αυτό είναι σημαντική και η οικονομική τους ανάπτυξη και ευρωστία. Γιατί πολλές φορές το καλύτερο όχημα για, τη για την συμφιλίωση των λαών είναι η επικοινωνία και η εκπαίδευση. Και εδώ... Κυρία Κώστα. Ναι, είναι εξαιρετικό σημείο κίνηση η γνωμοδότηση για να συστήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό και για τη δική μα την Επιτροπή θέμα για την διασυνεργειακή συνεργασία, ιδιαίτερα στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Θα ήθελα να πω ένα-δύο πράγματα για τα όσα έχετε εντοπίσει στη γνωμοδότησή σα. Καταρχά, όταν μιλούμε για γραφειοκρατικές αρχές πρέπει να είμαστε πιο ακριβείς νομίζω γιατί μιλούμε για ένα θέμα θεσμικό το οποίο έχει να κάνει με τις διάφορες αρμοδιότητες, κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών στις διάφορες περιφέρειες γιατί υπάρχουν και αυτόνομες ε, διοικητικά περιφέρειες σε ορισμένες χώρες. Κάποιες άλλες να μην έχουν τέτοιου είδους ε, αυτονομία στην περιφερειακή τους οργάνωση οπότε ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε για διοικητική συνεργασία. Επίσης ε, θα πρέπει να αποτρέψουμε ένα κίνδυνο που ενδεχομένω να υπάρχει, το Ιντερεκ να μετατραπεί σε ένα ε, μοχλό ο οποίος μπορεί να δίνει κάποιους πόρους χωρίς όμως πραγματικά να ενισχύει μια γνήσια συνεργασία. Πρέπει να δώσουμε έμφαση ιδιαίτερα στη συνεργασία, να μην πηγαίνουν χρήματα αν δεν υπάρχει πραγματική συνεργασία. Στη συνέχεια θα ήθελα να πω ότι πρέπει να είναι ιδιαίτερα να είναι διασυνοριακός ο σχεδιασμός και η συνεργασία. Και τελευταίο, κινητικότητα στον χώρο της καλλιτεχνικής παραγωγής ε, και του πολιτισμού. Νομίζω ότι μπορούμε να μιλούμε για ένα artistic mobility, για μια κινητικότητα καλλιτεχνική ε, σε περιοχές που έχουν κάνει μεγάλες προβολές καλλιτεχνικού έργου στον χώρο του Interreg, που όμως έχουν μείνει μέσα στις δομές, δηλαδή στην κληρονομιά και πολύ λιγότερο στη συνεργασία, γλωσσία, διάλογο, ε, ζωντανές ε, παραστάσεις στις, ε, στα performing acts κτλ. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία πιστεύω γιατί πρέπει να μάθουμε να μεγαλώνουμε, να ζούμε μαζί. Και ένα τελευταίο είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι στον προσεχή προγραμματισμό, να υπάρχει στον προσεχή προγραμματισμό ενίσχυση αυτό που θα είναι τελικά το μεγάλο κομμάτι των περιφερειακών διαρθρωτικών ταμείων, ώστε στην διασυνοριακή αυτή συνεργασία να δοθεί μεγαλύτερη ενίσχυση για τα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά έργα. Αυτό για να προκαταλάβω λίγο και τη γνωμοδότηση για τα περιφερειακά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γουότς. Ε, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα, λέει η κυρία Ward, ιδιαίτερα λόγω της κατάστασης με τα σύνορα στην Ιρλανδία. Ε, ήμουν δύο μέρες επίσκεψη στη Βόρεια Ιρλανδία και πήγα στο Νιούρι, είδα εκπρόσωπους ε, επιχειρήσεων και από τα, τη βόρεια πλευρά και από την νότια πλευρά των συνόρων. Ε, υπάρχουν εκεί μια σειρά από κτίρια, κτηριακές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις ε, ε, που χρηματοδοτήθηκαν κατά 95% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόλις 5%, 5 δηλαδή της χρηματοδότησης προέρχεται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, χαιρόμαστε λοιπόν που το Ηνωμένο Βασίλειο αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν, να δημιουργείται πολιτική συνοχή και οικονομική συνοχή σε δύσκολες περιοχές Εάν το δούμε αυτό στα, στο πλαίσιο τώρα της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, ε, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που πάνε στο σχολείο ε, από τη μία πλευρά των συνόρων και ζουν στην άλλη. Και κάποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν απελπιστεί, κλαίνε. Δεν ξέρουν αν θα συνεχίσουν να πηγαίνουν τα παιδιά αυτά στο σχολείο με τους μαθητές τους. Και επίσης η Βόρεια Ιρλανδία ψήφισε την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου και γενικότερα οι νέοι ψήφισαν την παραμονή του Ηνωμένο Βασίλειου. Υπάρχει όμως και ένα άλλο ζήτημα για, που αφορά τους φοιτητέ ε, και την ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ε, Ορισμένε φορές μπορούν να θέλουν να πάνε από το βόρειο μέρος των συνόρων προ το Δουβλίνο ή από την Δημοκρατία της Ιρλανδίας ε, ε, για κάποια μαθήματα στη Βόρεια Ιρλανδία. Ε, συνάντησα λοιπόν ε, και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Belfast και θα ήταν καλό να σας κάνουμε μια αναφορά για τα ζητήματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γραμματικάκης έχει το λόγο. Ε, δεν θέλω να επαναλάβω όσα είπαν οι προηγούμενοι, αλλά να τονίσω ένα ιδιαίτερο παράγοντα που είναι η κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο νομίζω προγράμματα διασυνοριακά που απευθύνονται περισσότερο προς τις ε, έτσι αγνοημένες περιοχές της κάθε χώρας είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Γι' αυτό και θέλω να επενέσω την έκθεση του κυρίου Ζαγοράκη, διότι εμφανίζεται πλήρης, δίδει μεγάλη σημασία στα πολιτισμικά προβλήματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό εν ώψη και της μεταναστευτικής λέλαπας που ζουν ορισμένε χώρες, με την καλή έννοια το λέω, ε, και επίσης ε, προσπαθεί να προλάβει αδυναμίες που έχουν φανεί από το παρελθόν κυρίως γραφειοκρατικές αδυναμίες. Είμαι λοιπόν πολύ αισιόδοξο ότι χάρη στην έκθεση του κυρίου Ζαγοράκη θα κάνουμε ακόμα ένα βήμα μπροστά σε αυτό το τεράστιο θέμα για πολλές χώρες και που θα ευνοήσει την πορεία προς ένα καλύτερο μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Θέλω να προσθέσω σε αυτό που είπε η κυρία Κώστα. Εξ όσων γνωρίζω, στα προγράμματα Interreg δεν προωθούνται εθνικά προγράμματα, αλλά μόνο συνεργατικά προγράμματα, τα οποία πρέπει να σχεδιάζονται για από κοινού. Αυτό είναι κατοχυρωμένο στο πλαίσιο και στο καθεστώς αυτών των προγραμμάτων Interreg. Θέλω να το τονίσω αυτό. Στα προγράμματα Interreg η συνεργασία λειτουργεί πολύ ε, καλά τα χρηματοδοτικά μέσα ε, είναι αυτά που λείπουν και γι' αυτό πρέπει πάντοτε να μοιράζονται ανάμεσα σε, σε έργα υποδομή, σε έργα εκπαιδευτικά ε, κτλ. Θέλω απλά να διευκρινίσω. Ναι, το πρόβλημα είναι το εξής. Ακριβώς αυτό ζητώ και εγώ. Έτσι πρέπει να είναι. Αλλά έχοντα και την εμπειρία περιφερειακή διοίκηση διαχείριση, το έχω επιδιώξει μάλιστα. Αλλά, αλλά υπάρχουν κάποιοι φραγμοί ε, γραφειοκρατικοί μεταξύ των διοικητικών αρχών που δεν επιτρέπουν τη δυνατότητα όχι του σχεδιασμού, αλλά τη πραγματική συνεργασία. Και τελικά ο καθένα προχωράει από την πλευρά του. Το λέω όχι ω στόχο, το λέω ω πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό πρέπει να γίνεται πολύ σοβαρή αξιολόγηση των προγραμμάτων αυτών, ώστε να είναι γνήσια υπερσυνοριακά, Όχι δύο χώρε που συνεννοούνται, κάνουν την πρόταση και μετά ο καθένα ε, στη γωνιά του κάνει το μέρο τη δουλειά που του αναλογεί. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μπέλτ. Ναι, συγγνώμη, άργησα να ζητήσω το λόγο προηγουμένω. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του. Ε, θα ήθελα να αναφερθώ καταρχήν στην ανακοίνωση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πριν περάσω στο πολιτιστικό σκέλος. Προέρχομαι από μια πολύ μεγάλη περιοχή διασυνοριακή, τη Λορένη, όπου ένας στους δέκα εργαζόμενους ε, διασχίζει τα σύνορα. Είναι προφανές ότι οι διασυνοριακές περιοχές, οι παραμεθόριες, ε, αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες οικονομικές δυσκολίες ε, και υπάρχουν επίσης σημαντικές ανισότητες. Ο μέσος μισθός είναι 3.709 ευρώ στο Λουξεμβούργο και 2.600 στη Λορένη, όπου βέβαια και η ενεργεία είναι υψηλότερη από τον Γαλλικό Μεσόρο. Μπορούμε να μιλάμε για κινητικότητα και για σύμπραξη ε, για την κατάρτιση όταν είναι σαφές ότι η ροή θα είναι προς τη μία μόνο κατεύθυνση. Ε, βεβαίως μπορεί αυτό να βοηθήσει στο να μειωθεί η ανεργία στη Λορένη, αλλά εδώ και 20 χρόνια όλο και αυξάνεται το ποσοστό των διασυνοριακών εργαζομένων χωρίς αυτό να οδηγεί σε θετικό αντίκτυπο για την οικονομία. Απλά ε, έχει αυξηθεί ε, η τιμή των ακινήτων και υπάρχουν κάποια φορολογικά έσοδα. Επίσης αυξάνονται οι ανισότητες εντός των ίδιων των περιοχών και οι τοπικές, ε, ο τοπικός πληθυσμός δημιουργεί, αρχίζει μάλλον ε, να νιώθει άσχημα, όπως στην Ελβετία. Χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις ό,τι αφορά τις υποδομές. Όταν ζητούμε λοιπόν διαπεριφερειακή συνεργασία, καλά κάνουμε, αλλά είναι δύσκολη εφαρμογή. Παραδείγματο χάρη, η ανατολική περιοχή ε, της ε, Γαλλίας δυσκολεύεται να τα βρει με το Λουξεμβούργο σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση ενός νέου ε, κομματιού αυτοκινητόδρομου που κοστίζει 1,3 με 1,6 δις και που είναι απαραίτητο αυτό το κομμάτι του κινητόδρομου ε, έχουμε 40-50 λεπτά καθυστέρηση στο δρόμο χωρίς αυτό το κομμάτι υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα με το Λουξεμβούργο φορολογικό βέβαια διότι το Λουξεμβούργο θέλει όσοι εργάζονται εκεί να πληρώνουν τον φόρο τους εκεί και τα λοιπά δεν έχω άλλο χρόνο νομίζω έτσι Ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Σύντομα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μια σύντομη παρέμβαση. Θα ήθελα να καλωσορίσω το κείμενο του εισηγητή ε, και την υποστήριξη της Επιτροπής Πολιτισμού προς την ανακοίνωση. Γενικότερα σημειώσαμε όλα όσα υπόθηκαν και θα διαπιστώσετε ότι στα νέα προγράμματα Interreg που θα ξεκινήσουν το 2021 ε, θα συνεχίσουμε να επενδύουμε ιδιαίτερα σε ζητήματα πολυγλωσσίας, ε, σε πολιτιστικές δραστηριότητες. Ε, εμείς από πλευράς Κομισιόν σίγουρα θα δώσουμε όθηση σε αυτό. Βεβαίως τα προγράμματα είναι στα χέρια των εταίρων μας, διασυνοριακό επίπεδο. Εμείς διαπραγματευόμαστε μαζί τους. Η απόφαση όμως θα πάρθει από τις αρμόδιες αρχές, ε, τις εμπλεκόμενες αρχές. Ε, η Γενική Διεύθυνση Ρίτζιο έχει συντάξει αυτή την ανακοίνωση, διότι εμείς ασχολούμαστε με τις διάφορες ε, περιφέρειες, ε, όμως ήταν μια διεπηρεσιακή προσπάθεια, κοινή, συμμετείχε η Γενική Διεύθυνση Παιδείας και συνεργαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε την υποστήριξη για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητε διασυνοριακά. Παραδείγματο χάρη η πρωτοβουλία για το σήμα το γλωσσικό που δίνει έμφαση στην αναγνώριση και στην προώθηση των προσπαθειών πολυγλωσσίας ε, διασυνοριακά. Το θέμα των δεξιοτήτων επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εκεί πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά πράγματα. Τα κράτη-μέλη ε, έχουν μεγάλη ευθύνη εδώ έτσι ώστε να είναι πιο εύκολα και πιο συστηματικά αυτά τα πράγματα. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ των χωρών Benelux ε, που έχει περάσει τώρα σε νέα παρθένα εδάφη ε, μιας και αναγνωρίζονται πλέον δεξιότητες και προσόντα μεταξύ των τριών αυτών χωρών, Λουξεμβούργο, Βέλγιο, κάτω de facto, εξάντε δηλαδή, εκ των προτέρων, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κάποια διαδικασία. Ε, σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτές τις καλές πρακτικές τι οποίες ανακαλύψαμε και εμεί θα συνεχίσουμε να προωθούμε ε, την πολυγλωσία και τις πολιτιστικέ δραστηριότητε διασυνοριακά. Ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε και για αυτήν την εξαγγελία της περαιτέρω ανάπτυξης και διεύρυνσης των προγραμμάτων Interreg. Είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι η Κομισιόν ανεξάρτητα από τον τομέα πολιτικής καταφέρνει και συντονίζει τις υπηρεσίες της, υπάρχει καλή συνεργασία. Θα παρακολουθούμε και εμείς βεβαίως αυτή τη διαδικασία συστηματικά και θα συντάξουμε και γνωμοδότηση ως Επιτροπή Πολιτισμού. Θέλω, κλείνοντας, να ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Ζαβοράκη να πω όμως πριν το κάνω αυτό ότι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών είναι 22 Μαΐου και η ψηφοφορία θα γίνει στις 19 Ιουνίου. Κύριε Ζαγοράκη, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Όσο πιο σύντομα μπορείτε. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από αυτό που έχουμε ακούσει. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συναδέλφους για τα πολύτιμα σχόλιά τους και να είστε σίγουροι όλοι ότι με τη συνεργασία που θα έχουμε τα αποτελέσματα θα είναι επιθυμητά και αυτό που θέλουμε γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Κάθε επιτυχία στο έργο σας και θα επανέλθουμε βέβαια στο θέμα αυτό. Και περνάμε στο σημείο 6 σημερινή σα διάταξη και θέλω να ζητήσω από του δύο προσκεκλημένου μα να έρθουν στο βήμα. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την ε, εφαρμογή ε, τη, του, την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτικής Κληρονομιάς. Μια στιγμή, να μπορέσουν όλοι να καθίσουν. want to Thank you very much. I put it here. So, jetzt haben wir auch den richtigen Rahmen geschaffen. Λοιπόν, ωραία. Είμαστε πλαισιωμένοι πλέον και περνάμε στην ανταλλαγή απόψεων. Βρισκόμαστε στο μέσο ε, αυτού του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς και γι' αυτό είναι ιδιαίτερη χαρά μου που έχουμε σήμερα μαζί μας τους εκπροσώπους της Κομισιόν για να συζητήσουμε το τι συνέβη στο, τους προηγούμενους μήνες και τι σχεδιάζεται να γίνει ε, μέχρι το τέλος του 2018. Καλώς ορίζω λοιπόν την Κατρίν Μανιά που είναι η επικεφαλής της ομάδας για το ευρωπαϊκό έτος καθώς και τον κύριο Μισελ ε, Μανιέ που είναι διευθυντής για πολιτική πολιτική στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λίγο χρόνο δυστυχώς έχουμε. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αφιερώσουμε και λίγο χρόνο στη συζήτηση θα σας παρακαλούσα να περιορίσετε τις παρουσιάσεις σας στα 15 λεπτά συνολικά. Πώς θα τα μοιράσετε είναι δικό σας θέμα. Σας δίνω το λόγο. 15 λεπτά έχετε. Κύριε Μανιέ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω ε, την ε, Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την πρόσκληση, αλλά και για την υποστήριξη, τη συνεχή υποστήριξη που είχαμε από την αρχή αυτής της κοινή περιπέτειας. Είναι λοιπόν μια ευκαιρία σήμερα να σας ε, δώσω μια πρώτη αναφορά για αυτό το έτος. Διάβασα ξανά την νομική βάση μας πριν έρθω και διαπίστωσα ότι Είμαστε ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους μας, ε, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης ε, λειτουργούν. Ε, όπως ξέρετε, η χρονιά ξεκίνησε επισήμως στις 7 Δεκεμβρίου πέρυσι στο Φόρουμ Πολιτισμού που οργανώθηκε στο Μιλάνο και είχαμε μια σειρά από εκδηλώσεις που έδωσαν τον ακτήριο Λάκτης μας το έτος σε πολλά κράτη-μέλη. Είχαμε τρεις συναντήσεις των Εθνικών Συντονιστών και των Εμπλεκομένων Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών το 2017 και άλλη μία το Μάρτιο φέτος. Οι επόμενε συναντήσει θα λάβουν χώρα τον Ιούνιο στι Βρυξέλλες και τον Νοέμβριο στο Λάιπτσιχ, στη Λιψία, στα πλαίσια της Denkmalfair. Το κοινοβούλιο που συμμετέχει σε αυτές τις συνεδριάσεις ε, θα διαπίστωσε ότι υπάρχει ενθουσιασμό ότι λειτουργεί καλά, ε, λειτουργήσαν καλά αυτές τις συνεδριάσεις, ε, προχωράει η εκστρατεία σύμφωνα με το πρόγραμμα και πολλά μέσα ενημέρωση εθνικά αλλά και τοπικά ε, τονίζουν αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Κληρονομιάς ε, και το hashtag μας προχωράει στα κοινωνικά δίκτυα. Ήδη ε, έχουμε δώσει το σήμα μας σε διάφορα project σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είτε αυτά είναι ευρωπαϊκά τα project, είτε πρόκειται για project τα οποία έχουν ξεκινήσει εθνικοί συντονιστές. προγράμματα συνεργασίας επίσης έχουν επιλεγεί μετά από μια έκκληση του, της Δημιουργικής Ευρώπης ε, ολοκληρώνεται η διαδικασία επιλογής. Μιλάμε για ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ περίπου που είχαμε προβλέψει για αυτό το σκοπό. Επίσης υπάρχουν και δράσεις επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο. Αυτή την εβδομάδα η αντιπροσωπεία μας στο Μεξικό, παραδείγματο χάρη, οργάνωσε μια εκδήλωση με εκατοντάδες ε, συμμετέχοντες Είχαμε και ένα άρθρο του New York Times για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Κληρονομιάς. Έγινε και μια εκδήλωση στην Κούβα. Όπως αντιλαμβάνεστε, το ευρωπαϊκό αυτό έτος ξεπερνάει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έχουμε μια πρώτη ευκαιρία να κάνουμε έναν απολογισμό ε, στην Σύνοδο Κορυφής για την κληρονομιά ε, στην, την εβδομάδα 18 Ιουλίου στο Βερολίνο. Το βασικό μου μήνυμα προς εσάς είναι ότι αυτό το έτος ήδη ε, παρουσιάζει τόσα ωφέλη που είναι σημαντικό να μην την αφήσουμε χωρίς συνέχεια. Το λογικό είναι όταν ολοκληρωθεί το έτος αυτό να μειωθεί το ενδιαφέρον και να ολοκληρωθούν απλώς κάποια project και να γίνουν και κάποιες εκθέσεις. Ε, γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείναμε τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την πολιτική κληρονομιά σύμφωνα με την ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθούν τα θεσμικά μας όργανα εδώ για κάποια χρόνια και που είναι ε, και στην βάση αυτού του ευρωπαϊκού έτους θέλουμε όλες οι δράσεις, όλες οι πολιτικές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο συνεισφέρουν στην διαφύλαξη και στην αξιοποίηση του, της προσοχής κληρονομιάς θέλουμε να συγκεραστούν. Αυτή η πρόταση είναι την, προέρχεται από τον Επίτροπο Ναύρατσιτ, που οργάνωσε, σε μια συνεδρία που οργάνωσε στο Πλόβντιβ στην ε, Φιλιππούπολη η Βουλγαρική Προεδρία και αναφέρεται αυτό και στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τον Πολιτισμό που θα εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτή η ιδέα ε, θα μεταφραστεί και σε συγκεκριμένε οικονομικέ προτάσει που προετοιμάζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα έτη 2021 έως 2027. Ελπίζουμε ε, να έχουμε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για άλλη μια φορά, έτσι ώστε αυτό το μεσομακροπρόθεσμο πρόγραμμα ε, να μπορέσει να ευοδοθεί, έτσι ώστε αυτή η σημαντική επένδυση που είχαμε αυτό το έτος να αποφέρει καρπούς. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην Κατρίν, αν δεν έχετε αντίρρηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ Μισελ. Ε, καλημέρα σε όλες και όλους. Θα προσπαθήσω τώρα να σας δείξω κάποιες εικόνες και να σας δώσω και κάποια αριθμητικά στοιχεία για να συμπληρώσω την παρουσίαση. Έχουμε, σας έχουμε μοιράσει νομίζω αυτή την παρουσίαση PowerPoint επειδή έχουμε λίγο χρόνο και θέλουμε να υπάρξει μια δυνατότητα ανταλλαγή απόψεων. Δεν θα σας παρουσιάσω όλες αυτές τις διαφάνεις ε, ε, προφορικά. Τις βλέπετε πάντως μπροστά σας. Θα ήθελα εν συντομία να αναφερθώ σε κάποια παραδείγματα εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτου, ε, να σα δώσω κάποιε πληροφορίε ε, για την ε, επικοινωνιακή μας καμπάνια και να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Έτο δεν αφορά μόνο την επικοινωνία ούτε τι εκδηλώσει. είναι και μια επένδυση σε συγκεκριμένα προγράμματα, σε συγκεκριμένε ευρωπαϊκέ πρωτοβουλίε που θα μα επιτρέψουν να οικοδομήσουμε βιώσιμα πέρα από το έτος 2018 αυτό, αυτή την προσπάθεια. Ε, οι εκδηλώσεις πρώτα. Είχαμε περίπου 100 εκδηλώσεις ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο υπάρχουν όπως ξέρετε εθνικοί συντονιστές σε κάθε χώρα οι οποίοι είναι εξαιρετικά δραστήριοι και ως τώρα έχουμε 2.300 εκδηλώσεις στα κράτη-μέλη που έχουν αυτό το σήμα, αυτό το label του ευρωπαϊκού έτους που αφορούν περίπου ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Αν δούμε αυτά τα στοιχεία, τα προβάλλουμε ε, στο σύνολο του έτους και αν συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό θα φτάσουμε στα 8.200, στις 8.200 εκδηλώσεις στο σύνολο τη Ευρώπη. Όλα αυτά βεβαίω μπορείτε να τα βρείτε και στην ιστοσελίδα μα, όπω είπε ο Μισελ, ε, το έτο. Ε, ξεκίνησε στι 7 Δεκεμβρίου στο Μιλάνο, ήταν η κυρία Καμερτέβερ, το κύριο Σταγιάννη, ε, είχαμε και εθνικέ εναρκτήριε εκδηλώσει, σε πολλά κράτη-μέλη. Να εδώ ένα κατάλογος μαζί με κάποιε εικόνε, Βλέπετε μια εικόνα ε, στις 31 Ιανουαρίου στο, στις Βρυξέλλες ε, με την προβολή πάνω στο Δημαρχείο ε, ήταν 8 επίτροποι μαζί με τον κύριο Γιούνκερ εκείνη τη μέρα στο Δημαρχείο των Βρυξελών να σας δείξω τώρα και κάποια, κάποιες εικόνες από τις εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στις Βρυξέλλες έχουμε περίπου μία διάσκεψη το χρόνο εδώ βλέπετε τις αφήσει ε, των τελευταίων εκδηλώσεων, αλλά λαμβάνουν χώρα και εκδηλώσεις ε, σημαντικές τώρα, σύντομα, τον Ιούνιο, παραδείγματος χάρη ε, οργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο μια εκδήλωση για τους νέους. Θα έχουμε εμείς εκεί ένα περίπτερο για το Ευρωπαϊκό Έτος και θα παρέμβουμε, συμμετέχουν χιλιάδες νέοι από όλη την Ευρώπη και χαιρόμαστε που θα συμμετάσχουμε. Μια άλλη σημαντική στιγμή του Ευρωπαϊκού έτους ε, θα είναι η, η εβδομάδα 18-24 Ιουνίου στο Βερολίνο όπου η, η οργάνωση Europa Nostra ε, σε συντονισμό με τον εθνικό συντονιστή της Γερμανίας για το Ευρωπαϊκό Έτος οργανώνουν μια πολύ σημαντική σειρά εκδηλώσεων πάνω από 70 εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα εκείνη την εβδομάδα και που θα πληρωθούν μια πολύ σημαντική συζήτηση στις 22 Ιουνίου για το μέλλον του, της πολιτικής κληρονομιάς ε, στην Ευρώπη. Τώρα η, η επικοινωνιακή μας καμπάνια. Έχουμε και ένα βίντεο σε 24 γλώσσες ε, που μιλάει για αυτό το ευρωπαϊκό έτος. Ελπίζω να έχουμε τη δυνατότητα και τον χρόνο να σας το δείξουμε. Μια ιστοσελίδα και στις 24 γλώσσες ε, της Ένωσης ένα εξαμηνιαίο δελτίο τύπου ε, με πάνω από 6.000 ε, συνδρομητές, ελπίζω να είστε και εσείς μεταξύ αυτών. Υπάρχει το hashtag, έχουμε, παροχή, έχουμε παρουσία μάλλον στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης. Έχετε λάβει και αυτό το φυλάδιο φαντάζομαι σε τρεις γλώσσες, υπάρχει και στις 24 γλώσσες, που θα φροντίσουμε να είναι διαθέσιμες αυτές οι μπροσούρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε πολύ ενεργοί στα κοινωνικά μέσα δικτύωση. Δεν θα σας διαβάσω τώρα όλα αυτά που βλέπετε στον κατάλογο. Ε, έχει ένα συγκεκριμένο, ρυθμό, έχουν ένα συγκεκριμένο ρυθμό τα κοινωνικά μέσα δικτύωση, οπότε πρέπει συνεχώς να κάνουμε κάτι καινούριο έτσι ώστε να μένει ζωντανό το ενδιαφέρον ιδιαίτερα των νέων που χρειάζονται γρήγορες αλλαγές και συχνές. Ο Μισελ αναφέρθηκε στο labeling, στο σήμα δηλαδή που δίνουμε σε κάποιες εκδηλώσεις, το σήμα το ευρωπαϊκό το οποίο χορηγούμε σε κάποιες εκδηλώσεις. Πάνω από 310 τέτοιες εκδηλώσεις ε, έχουν λάβει το σήμα μας ε, για τον, ως τον Απρίλιο, έτσι, οπότε θα έχουμε ακόμα περισσότερες. Ε, και είχαμε επίσης 2.700 700 ε, ε, πρωτοβουλίες, εκδηλώσεις, project τα οποία έλαβαν αυτό το σήμα σε εθνικό επίπεδο. Ε, εδώ βλέπετε κάποια παραδείγματα. Ε, στο αεροδρόμιο του Φιουμιτσίνο η αντιπροσωπεία μας στην Ιταλία εκεί ε, ετοίμασε αυτή την υπέροχη αφίσα που δείχνει τις ε, επενδύσεις των διαθροντικών ταμείων στην χώρα. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα. Ένα βιβλίο που έχει το σήμα, ένα βιβλίο χρωματισμού. Μου μένουν και λίγα λεπτά να αναφερθώ στα project ε, και στις πρωτοβουλίες που χρηματοδοτούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως είπα στην αρχή της παρουσίασης, εδώ είναι που ε, οικοδομούμε την κληρονομιά αυτού του έτους ε, για το μέλλον αυτού του έτους της Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς. Όπως ξέρετε έχουμε ένα προπολογισμό για χρηματοδότηση project ε, στα πλαίσια της Δημιουργικής Ευρώπης 5 εκατομμύρια ευρώ για αυτό το συγκεκριμένο συγκεκριμένο, συγκεκριμένο διαγωνισμό ας πούμε έπρεπε να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις χώρες για ποσά έως 200.000 ε, ευρώ ε, λάβαμε 60 project επιλέξιμα, είχαμε λάβει περισσότερα, αλλά 68 ήταν επιλέξιμα, που εκπροσωπούν 308 οργανώσεις στην Ευρώπη και επιλέξαμε 29. Δεν μπορώ ακόμα να σας παρουσιάσω τα project δυστυχώς, διότι μόλις ενημερώθηκαν οι, οι ενδιαφερόμενοι 25 Μαΐου Πάντως θα έχουμε την επίσημη ανακοίνωση, θα υπογράψουμε τις συμφωνίες χρηματοδότησης ε, με τους ενδιαφερόμενους ε, και βεβαίως θα πρέπει να ξεκινήσουν οι δράσεις από τον Ιανουάριο στο Σεπτέμβριο του 2018. Αυτή ήταν ε, απαραίτητη προϋπόθεση διότι πρέπει κάποιο ή μέρος του project να λαμβάνει χώρα εντός του ευρωπαϊκού έτους. Θα αναφερθώ τώρα στις 10 ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες που ανταποκρίνονται ε, σε τέσσερις στόχους και είναι η ραχοκοκαλιά της επένδυσής μας εδώ στο ευρωπαϊκό έτος. Ε, τέσσερις λοιπόν είναι οι πυλώνες, η δέσμευση, η βιωσιμότητα, η προστασία και η καινοτομία. Η κάθε μία από τις πρωτοβουλίες αυτές περιλαμβάνει πολλές δράσεις και κάθε μία από αυτές ανταποκρίνεται στους στόχους που είχαμε θέσει στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους στην απόφαση που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Για λόγους χρόνου βέβαια δεν μπορώ να αναφερθώ στην κάθε μία πρωτοβουλίε πρωτοβουλίες αυτές. Ε, εάν θεωρείτε ένα αναγκαίο βεβαίω μπορώ να το πράξω. Να σα δώσω, δώσω όμως κάποια παραδείγματα συγκεκριμένων δράσεων που έλαβαν χώρα στα πλαίσια αυτών των πρωτοβουλειών. Παραδείγματο χάρη για την πρώτη πρωτοβουλία είναι ο στόχος να συμμετάσχουν όσο γίνεται περισσότερο Ευρωπαίοι σε δράσεις που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή κληρονομιά ε, και τα άτομα με αναπηρία. Με την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης δημιουργήσαμε ένα βραβείο το οποίο θα επιβραβεύει τις πόλεις που έχουν κάνει κάτι ιδιαίτερο έτσι ώστε η πολιτική κληρονομιά είναι προσβάσιμη. Στις 4 Δεκεμβρίου θα απονεμηθεί αυτό το βραβείο στις Βρυξέλλες. Ένα άλλο παράδειγμα σε ό,τι αφορά την συμμετοχή των νέων. Έχουμε πολλές δράσεις που αφορούν τα σχολεία. Μία από αυτές είναι να έχουμε φέτος το, την πολιτική κληρονομιά ως θεματική για όλες ε, ε τις, ε, ε, τις διαδικασίες e-twinning της, μεταξύ σχολείων από διάφορες χώρες της Ευρώπης Δεν έχω πολύ χρόνο, οπότε δεν θα αναφερθώ σε κάθε μία από πρωτοβουλίε αυτέ. Θα φτάσω τώρα στις δύο τελευταίες διαφάνειες για να σας θυμίσω ότι προτείνουμε ήδη την, στα ε, πλαίσια της νέας ατζέντα για τον πολιτισμό που θα, που θα ανακοινωθεί σύντομα θα αναφέρει, να αναφέρει ένα σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή πολιτική και τα, δύο επόμενες σημαντικές ημερομηνίες για τις συναντήσεις που θα έχουμε τους εθνικούς συντενιστές του Ευρωπαϊκού έτους και την κοινωνία των πολιτών και τους πολιτιστικούς φορείς που μας συνοδεύουν δηλαδή στην υλοποίηση αυτού του έτους θα γίνουν στις Βρυξέλλες αρχές Ιουνίου η πέμπτη εξ αυτών και η τελευταία στη Λιψία αρχές Νοεμβρίου ε, παράλληλα με την ε, ε, με το Denkmal, το... την εκδήλωση για λοιπόν την πολιτική κληρονομιά την τοπική. Αυτά σε ό,τι αφορά την παρουσίασή μου. Δυστυχώ δεν μπορούσα να παρουσιάσω την κάθε μία από αυτέ τι διαφάνειε. Εάν θέλετε, εάν έχετε ερωτήσει, μπορώ να επανέλθω. Ευχαρίστω. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση και την όντως εντυπωσιακή ως προς το περιεχόμενο παρουσίαση. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και την διάσκεψη υψηλού επίπεδου που έχουμε κάνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που θα κάνουμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κατόπιν επιθυμίας που εξέφρασε και ο πρόεδρος Καταγιάννη και η Επιτροπή μας 26 Ιουνίου. Στο <clears throat> σημειώσετε παρακαλώ. Και για να προχωρήσουμε στη συζήτηση θα ακολουθήσουμε τη διαδικασία του πινκ-πονγκ που έχει αποδειχθεί πολύ χρήσιμη. Ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση και ξεκινώ με τη Σίλβια Κώστα. Σε παρακαλώ, στα δύο λεπτά. Ναι, ναι, πάρα πολύ ε, γρήγορα. Καταρχάς ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μανιό, αλλά και όλο το προσωπικό της ε, Γενικής Διεύθυνσης γιατί έκανε καταπληκτικές προσπάθειες ε, και νομίζω το αναγνωρίζουν και οι συνάδελφοι Διακόνου και άλλοι. Ε, βλέπουμε μια πάρα πολύ καλή διαχείριση με συμμετοχή των ενδιαφερομένων και χωρίς να θέλω να εξαντλήσω τώρα μια γενική αξιολόγηση, θέλω να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Πρώτον, η διαχείριση, η το governance και πιστεύουμε έχει πολύ μεγάλη σημασία να παραμείνει και αυτή η κληρονομιά από την χρονιά αυτή. Ε, πρέπει να παραμείνει δηλαδή ένα επίπεδο διαχείρισης σε διάφορα επίπεδα, γιατί είναι 13 οι γενικέ διευθύνσει που έχουν δραστηριοποιηθεί στην υπόθεση αυτή. Έτσι λοιπόν, ρωτώ, υπάρχει ένα σχεδιασμός, έχετε προγραμματίσει να διατηρήσετε αυτή τη διαχείριση, το governance. Δεύτερον, σε σχέση με τις άλλες γενικές διευθύνσεις, την ώρα που γίνονται και σχεδιάζονται τα πολυετή προγράμματα εσείς στην εμπειρία σας που σας επέτρεψε να συνεργαστείτε με άλλα προγράμματα του 2021-2027 μπορείτε να την αξιοποιήσετε και σε σχέση και με το Ταμείο Συνοχής για την πολιτιστική κληρονομιά γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό και υπόθηκε ήδη και από μια άλλη έκθεση ότι η δημιουργική Ευρώπη με 16 μόνο στην πολιτιστική κληρονομιά θα είναι δύσκολο να, και το υπόλοιπο τις δραστηριότητε, θα είναι δύσκολο να καλύψει όλε τι ανάγκε σα. Γι' αυτό ε, και η ψηφιακή και το. Και η DG Horizon και η DG Cult νομίζω ότι έχετε συνεργαστεί και διατηρείτε αυτόν τον διάλογο για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και τι βούλετε. Παρακαλώ κύριε Μανή. Ευχαριστώ. Ναι, πινκ πονγκ λοιπόν. Μια κυβέρνηση όντω. Θέλουμε να παραμείνει και μετά το 2018. Έχει δώσει πολύ καλά αποτελέσματα. Θα ήταν κρίμα να ε, μπει ένα τέρμα μετά το ε, εκπνοή της Ευρωπαϊκής Χρονιάς για τη συνοχή βεβαίως και θέλουμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τρόπο οικοδομητικό και αποτελεσματικό όπως εξ αρχής άλλωστε αυτή τη χρονιά από το, για το, το σχεδιασμό της χρονιάς. Θέλουμε να συνεχίσουμε ένα αποτελεσματικό διάλογο με τους αδέλφους και από τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακών Υποθέσεων για να διατηρηθεί η συνεχής αυτή προσήλωση και δέσμευση για την υποστήριξη της κληρονομιάς. Έξι δις έχουν από τα διαρθρωτικά ταμεία ε, χορηγηθεί έως το 2020 για την πολιτιστική κληρονομιά και ελπίζουμε στην προσοχή, του προσεχή προγραμματισμό να μπορέσουμε και να αυξήσουμε το μερίδιο αυτό. Ευχαριστώ κύριος Διακόνου. Ευχαριστώ. Δεν ε, έχω να πω κάτι συγκεκριμένο. Απλά να εκφράσω τη χαρά μου. Διότι στην αρχή της υλοποίησης αυτού του προγράμματος δεν περίμενα, πρέπει να σας πω ειλικρινά, ότι θα υπήρχε τόσο μεγάλη συμμετοχή ε, από πλευράς θεσμικών οργάνων. Γιατί συνήθως ο πολιτισμός δεν αποτελεί προτεραιότητα. Τώρα πια όμως είμαι πεπισμένος ότι με βάση και τα όσα ακούσαμε από τους εκπροσώπους της Κομισιόν, ότι η συμμετοχή αυτή και η προσήλυση είναι πάρα πολύ μεγάλη, εντυπωσιακή θα έλεγα. Εμείς ε, σε όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης είχαμε επιμείνει ε, στην, ε, στην ανάγκη να υπάρχει ενεργή παρουσία του Κοινοβουλίου σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις που διοργανώνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους. Γι' αυτό και θα ήθελα για άλλη μια φορά να καλέσω όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν σε αυτές τις εκδηλώσεις. Ευχαριστώ. Ε, μάλλον ε, τα συγχαρητήριά του σας εξέφρασε ο κύριος Διακόνου για, την, ε, για το έργο σας. Merci beaucoup, ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Διακόν. Βεβαίως και μας συγκινούν πολύ τα λόγια σας. Η υποστήριξη σας όμως είναι απαραίτητη για να, και για να λειτουργήσουν τα προγράμματα αυτά. Και αν αυτό το έχουμε καταφέρει είναι και χάρη στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των λοιπόν οργάνων και έτσι με μεγάλη υπερηφάνεια μπορούμε να το επισημαίνουμε αυτό γιατί έχουμε μπορέσει πέραν των φραγμών, των τείχων των ε, γενικών διευθύνσεων να εργαστούμε, να συνεργαστούμε έξι γενικέ διευθύνσει, αλλά ταυτόχρονα και να κάνουμε ένα σχεδιασμό για τη δράση αυτή για το ευρωπαϊκό έτο με διάφορα μέτρα, εκδηλώσει. Επίση, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έχει αποφασίσει όλε τι δημόσιε δραστηριότητε, διασκέψει με νέου κτλ. να τι αφιερώσει ε, στο έτο ε, Προστασία πολιτιστική κληρονομιά και με το Κοινοβούλιο βεβαίω έχουμε πολύ ε, καλή και έντονη συνεργασία. Πάντα βέβαια μπορούμε να τα καταφέρουμε και καλύτερα, αλλά ήδη είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και ευτυχεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τρίπλ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είχα την ευκαιρία εγώ να ηγηθώ το εις ε, εναρκτήρια εκδήλωση για το έτος πολιτιστική κληρονομιάς στο Αμβούργο. Άκουσα αρκετά επικριτικά όμως εκεί για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλω να σας ρωτήσω, ξέρετε ότι στα κράτη-μέλη πολύ συχνά παρουσιάζεται η, η εθνική διάσταση μόνο το τι έχει κάνει το... το κράτος με τις δομέ του και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ποτέ το Κοινοβούλιο. Γιατί αυτό συμβαίνει. Αλλά ε, χάρη σε εμά υπάρχουν όλα αυτά. Αλλιώ δεν θα υπήρχε το έτο πολιτιστική κληρονομιά και πρέπει να μεριμνείτε έτσι ώστε, να μεριμνάτε έτσι ώστε να παρουσιάσετε το κοινοβούλιο και η ε, συμβολή του. Και εγώ πλέον δεν είμαι να δεκτώ να παρασιωπάτε αυτό. Πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Και επίση, τι έχετε κάνει ώστε να διασυνδεθεί η φετινή χρονιά με το προσεχές έτος που είναι ευρωπαϊκές μάλλον με τις, ε, με, πρωτεύουσε τις ε, για το 2019. Έχετε κάνει κάποια διασύνδεση σε αυτό. Είχαμε κάπως συζητήσει και θέλω να δω αν υπάρχουν πιο συγκεκριμένα θέματα. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Για να συμπληρώσουμε αυτό για να συμπληρώσω αυτό που είπε και η Χέλγκα στην αρχή, εξ με μεγάλη δυσκολία πείσαμε την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ήταν καλή ιδέα ένα έτος πολιτιστικής κληρονομιάς γιατί η, ε, η, απάντηση, η που παίρναμε αρχικά ήταν ότι δεν έχει καμία σχέση με ανάπτυξη και απασχόληση και καλύτερα να το ξεχάσουμε. Άρα εμείς επιμείναμε και πολύ σωστά το είπε Σέλγα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αυτό που πίεζε πάντοτε και απαιτούσε να γίνει αυτή η χρονιά και με χαρά βλέπουμε τώρα ότι οι αρμόδιοι σε επίπεδο επεξεργασία των προγραμμάτων ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποδέχονται και βέβαια ε, αναλαμβάνουν τον συντονισμό των δραστηριοτήτων κτλ. Και τους υποστηρίζουμε, κύριε Μενή. Ναι, όντω. Ε, τέθηκε το θέμα της ορατότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι μας αφορά εμείς θέλουμε να είναι όσο γίνεται μεγαλύτερη η ορατότητα όλων των θεσμικών οργάνων που συμμετέχουν σε αυτό το project. Όσο περισσότερα θεσμικά όργανα θα έχουν δημοσιότητα και ορατότητα, τόσο περισσότερο το έτος αυτό θα φτάσει κοντά στους πολίτες. Και όπως είπε και η Κατρίν, εμείς αναγνωρίσαμε τον κρίσιμο ρόλο του Κοινοβουλίου ευθύ εξ αρχή σε αυτή την περιπέτεια. Είναι σημαντικό για μας αυτό, αν ορισμένες φορές δεν συνέβη, ε, αυτό είναι λυπηρό. Ξέρετε ότι έχουμε ορισμένε φορέ βέβαια περιορισμένε δυνατότητε παρέμβαση στι κυβερνήσει για να του βοηθήσουμε, να του ζητήσουμε να προβληθεί ο τάδε ή ο δίνα. Ε, σε ό,τι αφορά τι ε, πολιτικέ πρωτεύουσε, η εμπειρία μα έω τώρα δεν μα επιτρέπει να αξιολογήσουμε ακόμα τον ρόλο ε, τη ε, πολιτική κληρονομιά στι δύο αυτέ πρωτεύουσε. Ε, με αυτό το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράση όμω, εφόσον προκύψει, οι ευρωπαϊκές πολιτικές πρωτεύουσες σίγουρα θα παίξουν ένα ρόλο ε, για την κληρονομιά. Ε, ενδεχομένως θα πρέπει να συμμετέχει πιο καθαρά και πιο ορατά ε, το πολιτιστικό σκέλος ε, από κοινού με το σκέλος της πολιτικής κληρονομιάς. Ναι, θα ήθελα κυρία Τρίπελ να προτείνω και δύο συγκεκριμένες ε, δράσεις ε, για αυτό το θέμα της ορατότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε. 4 και 5 Ιουνίου, στη συνάντηση την επόμενη, όπως συνετέχουν όλοι οι εθνικοί συντονιστές μπορούμε να του θυμίσουμε τη σημασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κυρία Κώστα που είναι παρατηρήτρια εκεί, ε, μπορεί προφανώ να παρέμβει. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα είναι όλοι εκεί. Εκεί μπορούμε να τους θυμίσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θέλει να παρίσταται στις διάφορες εθνικές εκδηλώσεις. Και κάτι ακόμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε, και το απευθύνομαι βέβαια στο Κοινοβούλιο και πάλι, να δούμε εάν οι αντιπροσωπείε του Κοινοβουλίου σε διάφορα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν. Εμεί συνεργαζόμαστε πολύ με την αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής στα κράτη-μέλη. Ε, είναι αυτοί που μα βοηθούν στα πλαίσια ε, αυτή το της, α, αυτού ε, του ευρωπαϊκού έτου ε, στο Φιουμιτσίνο, η εικόνα που είδατε στο αεροδρόμιο προηγουμένω, το είναι δουλειά τη μόνιμη αντιπροσωπεία τη Κομισιόν εκεί. Ε, συνεργαζόμαστε πολύ μαζί του, του στέλνουμε πληροφορίε, οπότε είμαστε στη διάθεσή σα. Εάν ε, μα το επιτρέπετε, να έρθουμε σε επαφή με την αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα κράτη-μέλη. Σίγουρα είμαστε στη διάθεσή σα. Ευχαριστούμε πολύ καταρχάς για την υποστήριξη που μας παρέχετε και να επαναλάβω ότι εμείς θα έρθουμε σε επαφή και με τη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να δούμε μήπως ε, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να προβούμε σε κάποιες ενέργειες βελτίωσης ε, σε σχέση με το τι συμβαίνει τουλάχιστον μέχρι σήμερα. Ε, γιατί, εντάξει, έχει προκληθεί μια κάποια δυσαρέσκεια σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον το γεγονός ότι η δική μας υπηρεσία επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, θα μπορούσε σε κάποιες περιπτώσεις τουλάχιστον να είχε αναλάβει κάπως πιο ενεργή δράση. Προσεκτικά το διατυπώνω. Κύριε Όφλιν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καταρχάς να συγχαρώ την Κατρίν και τον Μισελ για αυτήν την περιεκτική παρουσίαση για το γεγονός ότι ε, έχουν ήδη διοργανωθεί ε, τόσες πολλές εκδηλώσεις φέτος. Δεν είναι έτος ε, ευρωπαϊκού πολιτισμού, αλλά πολιτιστικής κληρονομιάς. Και εγώ ε, ως ε, θεωρώ ότι η χριστιανοσύνη πρέπει να αναδειχθεί γιατί τα περισσότερα κτίρια μας, οι εκκλησίες, τα πανεπιστήμια, τα αναγεννησιακά κτίρια πραγματικά έχουν πάνω τους τη σφραγίδα της χριστιανικής θρησκείας. Και νομίζω ότι με κάποιον τρόπο υποβαθμίζεται αυτή η διάσταση, τουλάχιστον στις εκδηλώσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμησή μου ε, και επίσης ε, τα, τους επόμενους 7 μήνες προγραμματίζονται εκδηλώσεις οι οποίες θα αναδεικνύουν ακριβώς αυτή την χριστιανική διάσταση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Ποιος θέλει, λέει η Πρόεδρος, κύριε Μανιέ. Ναι, βεβαίως πάντα υπάρχει μια δυσκολία ε, να αγκαλιάσουμε το σύνολο του πλούτου μιας πολιτικής κληρονομιάς ε, επιμένοντας σε μία συνιστόσα. Βεβαίως, ε, η χριστιανική κληρονομιά αποτελεί μέρος ε, της ευρωπαϊκής πολιτικής κληρονομιάς και του έτους, αλλά δεν αναφέρεται αυτό ρητά στη νομική μας βάση, που αποτελούν ουσιαστικά τις γραμμές για, μένα, για Υπάρχουν βέβαια κάποιοι τομεί όπου αυτή η θρησκευτική διάσταση λαμβάνεται υπόψη, ενδεχομένω έμεσα. Μία από τι δέκα πρωτοβουλίε μα αφορά στην επαναχρησιμοποίηση των κτηρίων ε, πολιτική κληρονομιά. Σε πολλέ ε, χώρε ε, κάποια τέτοια κτηρία, συχνά θρησκευτικά κτηρία τεμένη, χάνουν τη λειτουργία τους στην κοινωνία, ερημώνονται. Θέλουμε λοιπόν από κοινού να εξετάσουμε πώς αυτά τα κτίρια, εκκλησίες ορισμένες, ορισμένα από αυτά, μπορούν να βρουν μια νέα κοινωνική λειτουργία, να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο χρήσιμο ε, για τις τοπικές κοινότητες και να προστατεύσουμε ταυτόχρονα και κάποια κτίρια τα οποία ιδάλλως θα εκλείψουν ή θα ε, υποστούν ζημιές. Λαμβάνεται λοιπόν, λοιπόν υπόψη αυτή η θρησκευτική κληρονομιά ε, Χωρί όμω να κοιτάζουμε προ το παρελθόν, κοιτάζοντα προ το μέλλον για να προσπαθήσουμε να του δώσουμε μια νέα διάσταση ε, στην σημερινή κοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σάντροβα. Ναι, ευχαριστώ για την παρουσίαση του Ευρωπαϊκού Έτους. Ε, παρουσίασα, ε, παρακολούθησα πολύ προσεκτικά όλες τις δραστηριότητες σας. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Διακόνου ε, εκτιμούμε ιδιαίτερα τη δουλειά σας να πω τώρα κάποια πράγματα πρώτα απ' όλα το χρονοδιάγραμμα για, την, ε, για το project και την ε, δημιουργική Ευρώπη θα είναι δύσκολο ιδιαίτερα για τις οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών της μη κερδοσκοπικές, οργανώσει οργανώσεις ε, να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα. Και λυπάμαι γι' αυτό. Θα δούμε τελικά τι θα συμβεί ε, βέβαια στις 25 Μαΐου όπως μας είπατε πάντως ε, ήταν δύσκολο να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις ένα ερώτημα Α, τώρα, ποια είναι η ορατότητα αυτού του έτους ε, εδώ στις Βρυξέλλες. διότι ξέρετε ότι υπάρχει ανταγωνισμός εδώ. Έχουμε το ευρωπαϊκό έτος του κινέζικου τουρισμού. Τέλος πάντων το τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Εδώ ε, στην πλατεία Σούμαν ε, υπάρχει μια μεγάλη αφίσα ε, που διαφημίζει αυτό το έτος, όμως ε, το ευρωπαϊκό έτος πολιτιστικής κληρονομιάς δεν είναι και τόσο ορατό στην πλατεία Σούμαν, ας πούμε. Ε, αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Μπορείτε να κάνετε κάτι γι' αυτό. Ευχαριστώ. Alors, sur le, le calendrier, euh, vous avez raison. Ναι, έχετε δίκιο για το χρονοδιάγραμμα. Μα έλειψαν έξι μήνε κατά την προπαρασκευή. Αργήσαμε λίγο, είναι προφανέ. Αυτή, η καθυστέρηση, αυτή την καθυστέρηση δεν μπορέσαμε να την ε, καλύψουμε πλήρω. Θα προτιμούσαμε να μπορούσαν να είχαν επιλεγεί αυτά τα project στην αρχή του έτους και όχι το Μάιο. Δεν μπορούσαμε όμως να κάνουμε κάτι άλλο. Αναγκαστήκαμε μάλιστα να συμπτύξουμε λίγο και το χρόνο που είχαν στη διάθεσή του αυτοί που έχουν υποβάλει τα project. Παρ' όλα αυτά πάντω υποστηρίξαμε πολύ καλά project. Θα το δείτε. Θα το δείτε. Αυτό είναι ένα καλό νέο. Τώρα για την ορατότητα στι Βρυξέλλες. Πρέπει να πω κυρία Σκόντροβα ότι πραγματικά εδώ αγγίξατε ένα σημείο που μας πονάει. Είναι πολλές εβδομάδες, πολλοί μήνες που ζητούμε ένα μπάνερ του ευρωπαϊκού έτους ε, στον Περλεμό. στον τοίχο του Περλεμό. Ε, δεν έχουμε λάβει θετική απάντηση. Αυτό δείχνει λοιπόν ε, ότι σε όλα τα θεσμικά όργανα έχουμε έτσι απογοητευτικές στιγμές με την Κυρική Δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω μιλήσει με όλο τον κόσμο. Θα του πω ότι έχουμε και τη στήριξη του Κοινοβουλίου, ε, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι περισσότερο από αυτό. Και εγώ λυπάμαι όσο και εσεί. Καλώ. Θα προσπαθήσουμε να τι στρώσουμε αυτέ τι Γενικέ Διευθύνσει Επικοινωνιακή Πολιτική. Κυρία award έχει τον λόγο. Θα συνεχίσω σε αυτό που έλεγε ο κύριος Φλίν η θρησκευτική κληρονομιά. Έχουμε πληθώρα δογμάτων και θρησκείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, είναι καθήκον μας να καταστήσουμε γνωστό και στις διάφορες οργανώσεις πιστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις ευκαιρίες που έχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχα παραδείγματι επικοινωνία με τον κύριο Μίλ που είναι ο ιδρυτής ε, του Ιδρύματος ε, Πολιτιστικ... Εβραϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς και δεν ήταν καν ενήμερος. Ένας άνθρωπος μόνος του βέβαια είναι, προσπαθεί να καταγράψει, κάνει αυτή την καταπληκτική δουλειά της καταγραφής, της χαρτογράφησης των συναγωγών της Ευρώπης και δεν ήταν καν ενήμερος και χαίρομαι ιδιαίτερος που μπόρεσα χάρη στη δική του τη δουλειά μπορέσαμε να οργανώσουμε ε, μια εκδήλωση για την εβραϊκή πολιτιστική κληρονομιά στην Κρακοβία φέτος με το Einbridge, το Διεθνές Ινστιτούτο ε, Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Ηνωμένου Βασιλείου, το Πανεπιστήμιο του Birmingham, το Πανεπιστήμιο της Κρακοβίας και άλλους φορείς. Πρέπει να ανασκουμποθούμε, πρέπει να δραστηριοποιηθούμε γιατί υπάρχουν δυνατότητες και ευκαιρίες στις χώρες μας για όλους αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν τόσα πράγματα και που έχουν μεγάλες ωραίες ιδέες. Ευχαριστώ πολύ κύριο Μανί. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Ward. Ε, είχα πει στον κύριο Φλίν, έχω δύο παραδείγματα να σας δώσω και αυτό ήταν ακριβώς το δεύτερο. Ε, το οποίο όμως ξέχασα να αναφέρω. Είναι πολύ σημαντική αυτή η αναφορά και η διάσκεψη στην Κρακοβία, στην οποία πρέπει να λάβουμε όλοι μέρος για να δείξουμε, να καταδείξουμε αυτή την πολιτιστική, θρησκευτική πολυμορφία και κληρονομιά. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ όχι μόνο για την παρουσία σας και παρουσίασή σας, αλλά και για τη συζήτηση. Ε, Εφτά μήνες μας μένουν περίπου, θα συνεργαστούμε όλοι μαζί για να σευθεί με επιτυχία όχι μόνο το έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά να του εξασφαλίσουμε και τη συνέχεια, την διάρκεια για την περίοδο από μετά το 2019 και μετά το 2019. Να μην χαθεί δηλαδή αυτό το ενδιαφέρον και η κινητοποίηση για την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά να διατηρηθεί και να συνεχιστεί και στο μέλλον. Ιδιαίτερα νομίζω ότι εδώ ήταν εύστοχο το σύνθημα «Where the past meets the future», εκεί που το παρελθόν συναντά το μέλλον. Νομίζω ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και για τη συνέχεια που θα δοθεί. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στη συνέχεια, στις διάφορες εκδηλώσεις σας, στα έργα, την ε, υλοποίηση αλλά και την παρακολούθησή τους. Και βεβαίως το θέμα αυτό εμάς θα μας απασχολήσει και στους προσεχείς μήνες. Υπενθύμησα ότι υπάρχει αυτή η διάσκεψη στις 26 Ιουνίου για μας και εμείς βεβαίως στο δεύτερο εξάμεινο έχουμε και μια κοινή εκδήλωση με τους εκπροσώπους των ε, Επιτροπών Πολιτισμού των Εθνικών Κοινοβουλίων σε μια διημερίδα εδώ στο Κοινοβούλιο που θα μας επιτρέψει να συζητήσουμε διδάγματα για το μέλλον και υλοποίηση προγραμμάτων και στο μέλλον με αποτελέσματα για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια για την πολιτιστική κληρονομιά και στο μέλλον. Ευχαριστώ λοιπόν και την κυρία Μανιάν και τον κύριο Μανιέ και εύχομαι κάθε επιτυχία. Merci. Λοιπόν, Παρακαλώ όλους όσοι δεν ανήκουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσοι μπορούν να μείνουν λοιπόν στην αίθουσα ευρωβουλευτές, βοηθοί, εργαζόμενοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμβουλοι. Όλοι οι άλλοι παρακαλώ να εγκαταλείψουν την αίθουσα γιατί προχωράμε σε συνεδρίαση και κλεισμένων των θυρών.